Κύριε Πρόεδρε μου, αξιότιμο μέλη του Κοινοβουλίου, θέλω να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την ευκαιρία που μου δώσατε να έλθω ενώπιόν σας στο σπίτι των λαών της Ευρώπης. Χαίρομαι που μπορέσαμε να συζητήσουμε θέματα τα οποία έχουν μεγάλη σημασία για τους Ευρωπαίους πολίτες. Τα θέματα της υγείας και της προστασίας των τροφίμων. Η Ευρώπη πρέπει να παίξει πρωτοπόρο ρόλο στον κόσμο σε όλους τους τομείς και σε αυτά περιλαμβάνονται και η υγεία, η ασφάλεια των τροφίμων. Μπορούμε λοιπόν με τον τρόπο αυτό να δείξουμε σε όλο τον κόσμο πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα παγκόσμια προβλήματα και τις παγκόσμιες προκλήσεις. Ως ιστορικός μπορώ να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η καλύτερη λύση για να προστατεύσουμε την ανθρωπότητα από τους πολέμους, από το μίσος και άλλες ασθένειες αυτού του είδους. Τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον υγειονομικό τομέα και την προστασία της ασφάλειας των τροφίμων είναι το καλύτερο παράδειγμα για τον κόσμο μας για να προστατεύσουμε την υγεία των ανθρώπων. Ως ε, πολιτικός μπορώ να πω ότι όλες οι πολιτικές παρατάξεις είναι ιδιαίτερα ταιριαστές για τις απόψεις τους όταν πρόκειται για τα θέματα της υγείας. Εγώ ως βουλευτής, ως ε, ένα άτομο που έχει σταθεί εκτοπισμένο στο παρελθόν του και έχει επανέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως υποψήφιος επίτροπος, όλα αυτά είναι πολύ συγκινητικά για μένα. Από τότε που ήμουν μικρός από τότε που έτρεχα στην τούντρα της Σιβηρίας ήθελα να φτάσω σε αυτή τη θέση που βρίσκομαι σήμερα. Εντάξει, πιο σοβαρά θέλω να σας πω ότι πάντα ονειρευόμουν ένα διαφορετικό κόσμο, ένα πιο λαμπρό κόσμο όπου θα μπορούσα να βοηθήσω τους ανθρώπους τους συνανθρώπους μου. Αυτό προσπάθησα να κάνω σε όλη μου τη ζωή. Αγαπητοί λοιπόν συνάδελφοι, αν συμφωνήσετε, εγώ θα μπορέσω να αφοσιωθώ ως επίτροπος στους ανθρώπους, στην υγεία τους, στην ευζωμία τους. Ένα πράγμα μπορώ να σας υποσχεθώ, θα εργαστώ σκληρά και θα συνεργαστώ μαζί σας και μαζί όλοι μπορούμε να το επιτύχουμε. Κάτι ακόμα θέλω να τονίσω. Έχουμε εδώ πέρα τη βίβλο μας, τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση το άρθρο 16 στην ένατη παραγραφό του λέει ότι η Προεδρία του Συμβουλίου θα ασκείται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών ε, με εναλλαγή σε επίπεδο ισότητας. Δική μου πρόταση ήταν αυτή στη συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης. Όλοι πρέπει να είναι σε επίπεδο ισότητος και όλοι πρέπει εξίσου να αγωνιστούν για τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Επίτροπε που απαντήσατε στις ερωτήσεις μας και που σεβαστήκατε και το χρόνο του πινκ-πονγκ που καμιά φορά είναι πολύ περιορισμένος διότι για κάποια θέματα χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος για να απαντήσει κανείς. Αυτοί είναι οι κανόνες στους οποίους κινούμεθα και τους κανόνες αυτούς σεβαστήκαμε κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Όπως σημειώσατε κι εσείς, Ανακοινώνω τη συνεδρίαση των συντονιστών θα λάβει η χώρα για την αξιολόγηση της ακροάσεως σήμερα ανάμεσα στις 3 και στις 4.30 το απόγευμα και κάποιοι συντονιστές θα κάνουμε την αξιολόγηση που αφορά την επίδοσή σας σήμερα στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ όλους για μια ακόμη φορά συνεργασία. Ζητώ συγγνώμη που χρησιμοποίησα το σφυράκι σε κάποιες φάσεις ήταν αναγκαίο για να μπορέσουμε να ε, παραμείνουμε εντός των χρονικών ορίων του κανονισμού. Ευχαριστώ και τα ξαναλέμε αργότερα.